Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να πάρετε τις θέσεις σας. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Τρεμόζα Ιμπαλσέης για την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2010. And uh, I would like to warmly welcome Θέλω εδώ να καλωσορίσω τον κύριο Μάριο Ντράγκη, ε, διοικητή της Ευρωπαϊκής Τραπέζης, Κεντρικής Τραπέζης και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία στο πολύ δύσκολο έργο που έχει αναλάβει. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τον εισηγητή μας, τον κύριο Τρεμόζα Ιμπαλτσέης, να λάβει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε Τράκη, σας καλωσορίζω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδεις, τους βοηθούς, ε, τους συμβούλους για την καλή συνεργασία που είχαμε για την εκπόνηση της έκθεσης αυτής. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα συζητάμε την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε στην Οικονομική Επιτροπή τον προηγούμενο μήνα. Όσον αφορά τη διαχείριση του χρέους, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την παρέμβαση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις αγορές. Και θέλω να τους ενθαρρύνω μέσα στις επόμενες εβδομάδες να συνεχίσουν με τις παρεμβάσεις τους οι οποίες έσωσαν το ευρώ. Χωρίς αυτές η κατάσταση σήμερα θα ήταν χειρότερη. Επίσης καταδικάζουμε τη, τους δισταγμούς για τη διαχείριση της κρίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις χώρες εκείνες οι οποίες δεν προχώρησαν σε μεταρρυθμίσεις. Πολλές φορές οδηγήθηκε γι' αυτό ακριβώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δράσει. Στην έκθεσή μα εκφράζουμε και τι ανησυχίε μα όσον αφορά τα όρια στην παρέμβαση Ευρωπαϊκή ε, Κεντρική Τράπεζα. Η νομισματική πολιτική δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Η κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για τη δικιά τη φορολογική και δημοσιονομική κατάσταση. Δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι στον ισολογισμό τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπάρχει μεγαλύτερη έκθεση σε κίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επί του παρόντος, είναι ο δανειστής, ο ίστατος δανειστής. Για τον τραπεζικό τομέα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ο ίστατος δανειστής από τον Μάιο του 2010. Έχει υπάρξει μια ροή πιστώσεων χωρίς όρια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς τις τράπεζες. Τράπεζε, οι οποίε αγοράζουν μεγαλύτερο, μεγάλο μέρο του χρέου, ε, από το δημόσιο χρέο. Η μαζική αυτή βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. θα ε, μπορούσε να αποτελέσει και κίνητρο όμως για καθυστερήσεις σε ορισμένες χώρες. Εμείς ψηφίσαμε ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης. Εγώ πιστεύω ότι η δημοσιονομική πειθαρχία αποτελεί προϋπόθεση για περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πιστεύω ότι η εθνική και ευρωπαϊκή προπολογισμοί είναι κάτι το οποίο πρέπει να τυχαίνει εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεσή μα επίση συμμεριζόμαστε την άποψη του κύριου Τρισέ, δηλαδή ότι χρειάζεται ένα Ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονομικών για να συντονίζει την οικονομική πολιτική των κρατών μελών και έτσι το ευρώ να είναι πιο αποτελεσματικό. Αυτή η κρίση χρέους δείχνεται σε μια νομισματική ένωση η δημοσιονομική πολιτική δεν είναι κάτι που μπορεί να παραμείνει αποκλειστικά στα χέρια των κρατών μελών. Επίσης, στην έκθεσή μας υπογραμμίζουμε ότι χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό σώμα το οποίο να ανακουφίσει κάπως την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το δημοσιονομικό της ρόλο και μέχρι τότε θέλουμε να δώσουμε ε, μεγαλύτερο ρόλο στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Κύριε Ντράγκη, ε, περιμένουμε τις δικές σας απόψεις για τις προτάσεις μας αυτές. Τέλος, όσον αφορά την διαφάνεια θέλω να έχουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Υπουργών Οικονομικών όπως γίνεται και στην Αμερική και στην Αγγλία και στην ε, Ιαπωνία και στην ε, Σουηδία της Τράπεζας των χωρών αυτών. Αλλιώς θεωρείται σαν σημάδι αδυναμίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θέλουμε ε, να γνωρίζουμε τα πάντα όσον αφορά τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Και γι' αυτό σήμερα θα ψηφίσουμε για τη δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ελπίζουμε να ακούσει τις δημοκρατικές φωνές του σώματος αυτού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, uh, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Τρεμόζα Ιμπαλσέης και τώρα κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε και ο εισηγήτης, ε, περιμένουμε με ανυπομονησία να μας πείτε ποιες είναι οι προτάσεις σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Τρεμόζα αξιότιμοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που κάνω την πρώτη μου εμφάνιση ενώπιόν σας με την ιδιότητα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2010. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να αποτίσω φόρο τιμή στον προκάτοχό μου, στον Jean-Claude Κατά τη διάρκεια της θητείας του, είχε έναν πάρα πολύ καρποφόρο και επικοδομητικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχω κάθε πρόθεση να ακολουθήσω τον δρόμο που χάραξε με την ίδια δύναμη, με την ίδια πυγμή ε, την οποία έδειξε. Η σημερινή μας σύνοδος είναι μια ευκαιρία για να ε, δούμε σφαιρικότερα τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, θα ήθελα να σχολιάσω και διάφορα γενικότερα θέματα που σχετίζονται με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας κάποια πράγματα για τις βασικές ε, πολιτικές, τα βασικά μέτρα μάλλον νομισματικής πολιτικής που αποφασίσαμε και εφαρμόσαμε το 2010 και 2011. Η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθοδηγείται από την ανάγκη εξασφάλισης της μεσοπρόθεσμης σταθερότητας στην Ευρωζώνη και σταθερότητα των τιμών. Αλλά αυτό είναι αμφίδρομο, έτσι το εννοώ. Δηλαδή, η σταθερότητα σχετίζεται και με τον προσδιορισμό των βασικών επιτοκίων και με την εφαρμογή μη πρότυπων μέτρων. Οι πιέσεις που διαπιστώνονται στις χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν ενταθεί με παράπλευρες αρνητικές συνέπειες ως προς την εμπιστοσύνη των αγορών. Ε, έχει αυξηθεί η δυνατότητα ύφεσης ως προς ε, τις χρηματοπιστωτικές ε, προοπτικές και παρατηρούμε αύξηση των πιέσεων ως προς τις τιμές και, την, και τα επιτόκια. Ε, και γι' αυτό το λόγο λάβαμε την απόφαση τον Νοέμβριο του 2011 να μειώσουμε κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες το βασικό μας επιτόκιο. Οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται σε διάφορες χώρες αποτελούν κόλλημα για την εφαρμογή της κοινή νομισματικής πολιτικής, διότι το πώς θα επηρεάσει αυτή η κοινή νομισματική πολιτική την πραγματική οικονομία είναι συνάρτηση της κατάστασης των ομολογιών ανακράτος μέλος. Ε, δηλαδή χρειαζόμαστε αποτελεσματικά μέσα για τη μεταφορά της νομισματικής πολιτικής προς την πραγματική οικονομία ε, πλήττονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις ε, διότι δεν έχουν επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. Και τώρα θα ήθελα να περάσω στα μη πρότυπα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα, τα οποία δεν μπορεί παρά να είναι περιορισμένα. Οι κυβερνήσει θα πρέπει μεμονωμένα και συλλογικά να αποκαταστήσουν την αξιοπιστία του ενώπιον των χρηματοπιστωτικών αγορών. Οι πιέσει στι αγορέ ομολογιών συνοδεύτηκαν από πιέσει στον τραπεζικό τομέα λόγω τη χρηματοπιστωτική διασύνδεση ανάμεσα στι κυβερνήσει και τις Τράπεζε. Η ΕΚΤΕ είχε αναλάβει διάφορα μέτρα και το 2010 και το 2011 για να με κατοχυρώσει ότι θα, την πρόσβαση μάλλον των τραπεζών στις πηγές χρηματοδότησης. Έτσι οι τράπεζες μπορούσαν να συνεχίσουν ε, την δανειοδότηση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η ΕΚΤ επέκτηνε την πολιτική της ούτως ώστε να εξασφαλίσει ε, ρευστότητα για τις τράπεζες ε, σε πάγια επιτόκια ε, με αντάλλαγμα εχέγγυα. Η αρχική εκπνοή των όλων των δράσεών μας που σχετίζονται με τη ρευστότητα αρχικά ήταν εξάμηνη και παρατάθηκε στους 12 ή και 13 μήνες. Έχουμε ένα νέο πρόγραμμα καλυμμένων ομολογιών, εξαγοράς καλυμμένων ομολογιών, 40 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, έχουμε προσφέρει προσφέρει περισσότερη ρευστότητα ως προς τα αμερικανικά δολάρια στις τράπεζες ε, για τρεις μήνες. Με συντονισμένη δράση για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, την Τράπεζα Ιαπωνίας, Τράπεζα της Αγγλίας, Τράπεζα Καναδά και Τράπεζα της Ελβετίας ε, έχουμε επεκτείνει τα μέτρα ρευστότητας ε, και έχουμε καλύψει διάφορες περιφέρειες της Ευρωζώνης. Επίσης, ως ε, κατεπήγον μέτρο αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε προσωρινές ρυθμίσεις ανταλα... διμερούς ανταλλαγής ρευστότητας, liquidity ε, swap, ούτως ώστε να υπάρχει επαρκής ρευστότητα για όλα τα νομίσματα εφόσον το υπαγορεύουν οι επιταγές ε, της αγοράς. Την ερχόμενη εβδομάδα την Πέμπτη θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ και είμαστε στην περίοδο προ των αποφάσεων. Δεν θα πρέπει λοιπόν να παρερμηνεύσετε αυτά που λέω και να προσπαθήσετε να μαντέψετε τι, πώς θα διαμορφωθούν μελλοντικέ νομισματικές ε, πολιτικές. Αλλά πραγματικά δοθεί στις κατάσταση δεν υπάρχουν και πολλά περισσότερα που θα είχα να προσθέσω τώρα σε σχέση με πρόσφατες δηλώσεις μου. Γνωρίζουμε τις πιέσεις που υπάρχουν λόγω των επισφαλών δημοσίων ομολογιών, τις πίεσεις που υπάρχει λόγω ε, των, ε, της έλλειψης πηγών χρηματοδότησης, ε, της έλλειψης επιλέξιμων εγγυήσεων σε κάποιους χρηματοπιστωτικούς τομείς. Γνωρίζουμε όλους τους κυκλικούς κινδύνους που σχετίζονται με την ύφεση, καθώς και όλες τις προκλήσεις που συνεπάγεται η αυξανόμενη ανάγκη κεφαλαίων για τις τράπεζες και για τις κυβερνήσεις. Θα ήθελα τώρα να περάσω στις προκλήσεις για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Το 2010 και 2011 είχε σημειωθεί σημαντική πρόοδος ως προς την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης. Αναγνωρίζω βεβαίως ότι αυτό δεν είναι προφανέ σε μεσούσε τη κρίση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη συμβάλει με αποφασιστικό τρόπο ε, στο να σημειωθεί αυτή η πρόοδο ε, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επικροτεί το έργο του Κοινοβουλίου. Το Six Pack στο περίφημο, δηλαδή η δέσμη των έξι οδηγιών, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, το Σύμφωνο Europlus, είναι πρωτοβουλίε ε, που έχουν προετοιμάσει το έδαφο, προλυάνει το έδαφο για στενότερο συντονισμό και εντονότερη εποπτεία των οικονομικών πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όλο λέει τη Ευρωζώνη. Παρ' Παρόλα αυτά ε, ε, διασχίζουμε μια πολύ δύσκολη φάση Έχουμε ήδη θεσπίσει νέους μηχανισμούς ε, και βλέπουμε κάποια θετικά αποτελέσματα, ε, αλλά ελάχιστα σε σχέση με την ε, αξιοπιστία των κρατικών δημοσιονομικών πολιτικών ενώπιον των αγορών. Επίσης, οι αλλαγές που γίνονται σε κυβερνητικό επίπεδο δεν έχουν ακόμη επηρεάσει δυστυχώς την επισφαλή θέση στην οποία έχουν περιέλθει χρηματοπιστωτικές αγορές. Άρα τίθενται θεμελιώδη ζητήματα και χρειαζόμαστε απαντήσεις. Στην καρδιά των ε, ερωτήσεων δεν είναι μόνο η αξιοπιστία των ε, κυβερνητικών πολιτικών ε, και αν θα εφαρμοστούν τα υπεσχημένα, αλλά είναι και ο κοινό σχεδιασμό τη μελλοντική δημοσιονομική μα διακυβέρνηση. Είμαι πεπισμένο ότι το νέο πλαίσιο εποπτεία θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία σύν το χρόνο και είμαι πεπισμένο ότι ακολουθούν τη σωστή τροχιά οι χώρε. Αλλά όμω χρειάζεται ένα, σημάδι αξιοπιστία, ώστε να έχουμε την ίστατη εγγύηση βράχει πρόθεσμα. Πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται η ΟΝΕ είναι μια νέα δημοσιονομική συμφωνία, δηλαδή μια θεμελιώδης δήλωση ε, των δημοσιονομικών κανόνων που ε, συνάμα με τις αμοιβέ δημοσιονομικές δεσμεύσεις ε, θα βοηθήσουν την Ευρωζώνη έχουμε μια συμφωνία που περιγράφει την ουσία της νομισματικής πολιτικής. Δηλαδή έχουμε μια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχουμε τον ενιαίο στόχο της διατήρησης της σταθερότητας των τιμών και γι' αυτό έλεγα ότι χάρη στη νέα δημοσιονομική συμφωνία θα μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε την πεντουσία των δημοσιονομικών μας κανόνων ε, και θα ε, ε, φροντίσουμε ούτω ώστε μεμονωμένα και συλλογικά να γίνουν πιο αξιόπιστες οι κυβερνητικές πολιτικές. Επαρκεί αυτή η νέα δημοσιονομική συμφωνία για να σταθεροποιηθούν οι αγορές. Μια αξιόπιστη μακροπρόθεσμη θεώρηση των πραγμάτων μπορεί να μας βοηθήσει βραχυπρόθεσμα. Αναρωτιόμαστε. Ε, λοιπόν, η απάντηση είναι ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο το πρώτο βήμα για να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία. Μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα στοιχεία, αλλά έχει σημασία η σειρά με την οποία προκύπτουν. Το πρώτο και πλέον σημαντικό είναι να καταλήξουμε σε αυτήν την νέα επίσημη συμφωνία η οποία ε, θα μας καλύπτει. Δηλαδή ε, υπάρχει θέμα αξιοπιστία αν ε, μακροπρόθεσμα ε, έχουμε θέσει τους στόχους μας. Ε, ε, είναι εξίσου σημαντικό για την επίτευξη αυτών των μακροπρόθεσμων στόχων να ξεκινήσουμε από την αξιοπιστία που πρέπει να κερδιθεί βράχη πρόθεσμα. Οι, επενδυτέ, οι επενδυτές, συγγνώμη, ούτως ή άλλως σε σχέση με τις κρατικές ομολογίες, ούτως ή άλλως παίρνουν μακροπρόθεσμες αποφάσεις. Χάρη στην Δημοσιονομική Συμφωνία επίσης θα περάσουμε ένα ηχηρό και επίκαιρο μήνυμα σε σχέση με την εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας στην Ευρώπη και θα χαράξουμε μια ξεκάθαρη πορεία για τη μελλοντική τη αν θέλετε, της Ευρωζώνης ε, για να πλαισιώσουμε τις ε, φιλοδοξίες των επενδυτών. Ε, ως προς τη νομική διαδικασία πιστεύω ότι θα πρέπει να αφήσουμε όλα τα σενάρια ανοιχτά. Δεν θα πρέπει να απορρίψουμε και την, το ενδεχόμενο τροποποίηση των συνθήκων, αλλά επίσης υπάρχουν και άλλα μέτρα, άλλες διαδικασίες πολύ ταχύτερες που πρέπει επίσης να εξετάσουμε. Ούτως ή άλλως οι επιχειρήσεις, οι οι αγορές και οι πολίτες περιμένουν από τους ε, ηθήνοντες Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσουν με αποφασιστικότητα για να εξέλθουμε από την κρίση. Χρειαζόμαστε θεσμούς, κανόνες και διαδικασίες που να είναι στο ύψος των απαιτήσεων μιας νομισματικής ένωσης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας, Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε μας δώσατε πολλά θέματα να σκεφτούμε και να σχολιάσουμε και τώρα ξεκινάει η συζήτηση και θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Γκάι Μίτσελ εν ονόματι του ΕΛΚ για δύο λεπτά. Κύριε, Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τον κύριο Γκντράγκη για την πρώτη του εμφάνιση εδώ ε, και για τις γρήγορες αντιδράσεις. Θέλω επίσης να χαιρετήσω την στήριξη της ΕΚΤ με ρευστότητα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την οποία δεν θα μπορούσαμε να έχουμε επιβιώσει. Αλλά έχουμε πολλά ερωτηματικά σε αυτό το σημαντικό σταυροδρόμι της ιστορίας μας και ε, ε, η ΕΚΤ πρέπει να είναι ο δανειστής τελευταίας διαφυγής. Τώρα, εάν θα πρέπει να είναι το EFSF ή η ΕΚΤ ή κάποιος άλλος μηχανισμός, αυτό δεν μας απασχολεί. Ε, αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι ότι αν χρειάζονται αλλαγές στις συνθήκες θα πρέπει να προχωρήσουμε με την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές σιγά σιγά θα υιοθετικούν διότι τέτοια επεξεργασία χρειάζεται χρόνο και ενδεχομένως θα χρειαστούν και δημοψηφίσματα και δεν νομίζω ότι έχουμε επαρκή χρόνο ε, και θεωρείται ότι είναι ε, νομική προϋπόθεση αλλά δεν μπορεί κανείς να λέει ότι θα γυρίσει πίσω ο Τιτανικός γιατί δεν δουλεύει ο σηματοδότης ε, και διότι εντωμεταξύ θα έχει χτυπήσει το παγόβονο και θα μαζεύουμε τα σπασμένα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει την ίδια πορεία όπως ο Τιτανικός και γι' αυτό υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία προηγούνται. Οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρέπει να κινηθούν τώρα. Είμαστε εξουσιοδοτημένοι, δεν είναι θέμα πολιτικών, είναι θέμα πολιτικών ανδρών και γυναικών και ελπίζω ότι θα είμαστε στο ύψος των περιστάσεων, διότι όλοι θα χρειαστεί να διαβάσουμε και να ξαναδιαβάσουμε ε, την ομιλία του Πολωνού Υπουργού προσφάτως στη Γερμανία, διότι καλό είναι είναι να κατανοήσουμε τι μας περιμένει για να εξασφαλίσουμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ο επόμενος είναι ο κύριος Κούτας για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε Ντάγκη, σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καταρχήν ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τρεμόζα για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε στην κατάρτιση αυτού του ψηφίσματος διότι στην κατάσταση ασταθείας η οποία υπάρχει ο λόγος της ΕΚΤ είναι πολύ σημαντική ε, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ε, ταραχές που διαδραματίζονται ή στις οικονομικές αγορές. Πρέπει να υπάρξει μια σταθερή πορεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης που πρέπει να μπορέσει να κινηθεί σαν χρηματοδότης τελευταίας διαφυγής εάν η τράπεζα αναλάβει αυτό τον κεντρικό ρόλο τότε θα υπάρξει μία αύξηση της εμπιστοσύνης σε όλη την Ευρωζώνη αλλά ο σημαντικός αυτός ρόλος της ΕΚΤ θα πρέπει να συμπληρωθεί με ριζικά μέτρα δηλαδή ενημέρωση των φορολογικών πολιτικών των κρατών μελών και ε, μία εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Σταθερότητος. Χαιρετίζω την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 23ης ε, δεκάτου όπου κηρύσσει ότι θα συσπηρωθούν τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να βρούμε μία αλληλέγγυη λύση πράγμα το οποίο θα μειώσει το κόστος του δανειοδοτήσεως και θα φέρει μεγαλύτερη ρευστότητα στις χρηματαγορές. Θέλω να πω κάτι ακόμη και ε, το πιστεύω ένθερμα ότι χωρίς μία κοινή φορολογική πολιτική δεν θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει στο μέλλον. Ευχαριστώ. Έχετε ε, δύο λεφτά τώρα κυρία Γκουλάρ. Κύριε Ντράγκη, ευχαριστώ. Χαιρόμαστε που σα βλέπουμε εδώ σήμερα και θα ήθελα να είχαμε και περισσότερους συναδέρφους εδώ μέσα στην αίθουσα για να τιμήσουν την παρουσία σα. Θέλω να μιλήσω για την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό ότι το υπενθύμησε η κυρία Μέρκελ, ο κύριο Μόντι και ο κύριο Σαρκοζή. Και εμεί, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούμε. Φυσικά η αρχή της ανεξαρτησίας σας δίνει μια παραπάνω ευθύνη εσάς και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όμως σας έχουμε εμπιστοσύνη για τις αποφάσεις που παίρνετε. Όλες οι σημερινές κερδοσκοπίες ε, μπορούν να πλήξουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά η εσωτερική σας οργάνωση με απασχολεί, που πιστεύω ότι πλήττει το ευρώ και την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θέλω όμως να επενθυμίσω και ένα άλλο θέμα, που είναι το θέμα της επικοινωνία. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να υπάρχει συζήτηση δεδομένου των πραγμάτων που διακυδεύονται. Είναι λογικό τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συζητάνε μεταξύ του έντονα. Όταν όμω λαμβάνονται αποφάσει, εγώ θα ήθελα συλλογικά να υπάρχει ένα ομαδικό πνεύμα και οι αποφάσει αυτέ να στηρίζονται προ όφελο ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι υπό εθνικό πνεύμα. Και θέλω και εγώ, όπως και το κοινοβούλιο μας εδώ, μεγάλη διαφάνεια. Το θέμα δεν είναι να διαβάζουμε τα πρακτικά, αλλά να μην περνάνε πράγματα στον τύπο και να μην ακούγονται από τα μέσα ενημέρωσης πράγματα, τα οποία να μην συμφωνούν τελικά με τόσα συλλογικά έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συνήθως λέμε ότι οι άντρες μιλάνε, ή, συγγνώμη, ότι οι γυναίκες μιλάνε πολύ. Σε αυτή την περίπτωση όμως φοβάμαι ότι οι άντρες θα έπρεπε να σιωπούν λίγο περισσότερο. Εμείς ε, πάντως ε, χαιρόμαστε για την ανακοίνωσή σας και θέλω να επιμείνω και σε κάτι ακόμα, ότι έχουμε μία συνθήκη, ένα νόμισμα και μία ανησυχία για πειθαρχία. Αυτή η ανησυχία για πειθαρχία πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και πρέπει να φροντίσετε να τηρείτε στο δικό σας ε, το αργότερο Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατά τα άλλα, σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ η κυρία Σουίνμπερν για ένα λεπτό παρακαλώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον πρόεδρο Ντράγκη για την ανάληψη των νέων καθηκόντων εν μέσω κυκλώνα. Ε, τώρα η καγκελάριος Μέρκελ και ο πρόεδρος Σαρκοζή και άλλοι έχουν δερμότερες συζητήσεις σε σχέση με τον νέο ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάνω απ' όλα η ανεξαρτησία ε, της ΕΚΤΕ θα πρέπει να κατοχυρωθεί κυρίως επειδή ε, διασχίζουμε μια κρίση. Είναι στοιχείο κλειδί. Αν ε, τα μέλη της Ευρωζώνης ε, θέλουν να είναι ο ίστατος δανειστής η ΕΚΤ θα πρέπει να νομιμοποιήσουν αυτό το ρόλο του και το ταχύτερο δυνατόν. Η ΕΚΤΕ δεν πρέπει να είναι πολιτικό ποδόσφαιρο και να δούμε ποιος θα, ποια κυβέρνηση θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Ε, τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα πρέπει να έχουν ένα προκαθορισμένο ρόλο, θα πρέπει να ε, βάλουν σε τάξη τα του οίκου τους, ε, τα κράτη-μέλη και δεν μιλάω μόνο για τα ε, μέλη της Ευρωζώνης. Έχουμε τη δέσμη των έξι οδηγιών ε, που εγκρίθηκε πριν από δύο συνόδους. Ε, καλούνται το ταχύτερο δυνατό να εφαρμόσουν τα μέτρα τα κράτη-μέλη και να τα προσαρμόσουν στις, στην εγχώρια κατάσταση για να μειωθεί το δημόσιο χρέος. Πραγματικά είναι στοιχείο κλειδί από η αξιοπιστία. Σας ευχαριστούμε κυρία Σουίνμπορν. Ο κύριος Χουντής τώρα. Έχετε ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Ντράγκη, ο καταστατικός στόχος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας για τη σταθερότητα των τιμών αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία μέσα σε αυτές τις συνθήκες αποδείχτηκε καταστροφικός. το υπογραμμίζει και η έκθεση δεν συμφωνώ προτείνω γίνεται η διασυζήτηση να αλλάξει ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας. δεύτερο το 2010 έκθεση την οποία συζητάμε η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα κρύφτηκε πίσω από τον πληθωρισμό με συνέπεια πρώτον να μην βάλει φρένο στην εκτείναξη των spreads δεύτερον να μην βάλει φρένο στη δράση τη μαφία των κερδοσκόπων των οίκων αξιολόγηση που του πέρασε και στο καταστατικό τρίτον να κρατήσει ψηλά το επιτόκιο εσεί το μειώσατε κατά το τελευταίο διάστημα σε περιόδου ύφεση πιο ψηλά από τι Ηνωμένε Πολιτείε, πιο ψηλά και από τη μεγάλη βρετανία. Τέλο, τα περί τη της ευρωπαϊκής κεντρικής είναι πολύ συζητήσιμα οι ανεξάρτητοι τραπεζίτες αγιοποιούνται σε σημείο πρωθυπουργοποίησης όπως έχουμε σε δύο χώρες επομένως χειραγωγείται πολιτικά και η κεντρική τράπεζα πρέπει να αλλάξει η σχέση αυτή πολιτικός κοινοβουλευτικός έλεγχος στην ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Um, Ευχαριστούμε κύριε Χουντή. Ο κύριος Μπλουμ τώρα. Έχετε ένα λεπτό κι εσείς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ελπίζω να μπορώ να σας λέω σύντροφο στις κατηδίαν συναντήσεις. Ε, τέλος πάντων, εγώ ήρθα, παρότι η προσέλευση είναι ιδιαίτερα ισχυρή σήμερα. Ε, ε, αντίθετα με τους συναδέλφους, ε, εγώ πιστεύω ότι το ενιαίο Δημόσιο Ταμείο, το ενιαίο Υπουργείο Οικονομικών και όλα τα σχετικά που προτείνουν οι συνάδελφοι είναι ένα μανιφέστο για μια ευρωπαϊκή δικτατορία ε, και ε, το συντηρητικό κόμμα φυσικά θα ανοίξει τις αγκάλες ε, και θα υποδεχτεί την πολιτική όπως κάνουν συνήθως και θα πουλήσουν ως δική τους αυτή την ιστορία στο Λονδίνο. θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν ποιητή ε, στον ε, πόλεμο που έλεγε ότι πρέπει, εν πάση περιπτώσει, πέρα από τα μέσα και τα όπλα και τα βέλη που έχεις να έχει και ένα στόχο, να ξέρει ποιον ε, στοχεύεις όταν πολεμάς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μέλτσερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, η έκτα ευθύνεται ε, για τη σταθερότητα του νομίσματος και από το 2010 έχει ε, δανείσει πέραν των 200 δισεκατομμυρίων στα καταχρεωμένα κράτη και έχει υπερβεί κατά αυτόν τον τρόπο την εντολή της. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η ΕΚΤ βρίσκεται σε μία ασαφή ζώνη μεταξύ της φορολογικής και της οικονομικής πολιτικής έχει χάσει την αξιοπιστία της και αυτό γίνεται εις βάρος Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στην κρίση δεν νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσει περισσότερο η ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διότι βρισκόμαστε ε, σε ε, πρόθυρα μίας καταρρεύσεως και μίας υφέσεως οπότε θα πρέπει ε, να μην συμπαρασύρει κανείς και τα ε, θερά κράτη της Ευρωζώνης στην καταστροφή. Ευχαριστώ και τώρα δίνω τον λόγο στους υπόλοιπους ομιλητές και πρώτα την κυρία Γκάλ Πέλτς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Γκράγκη στην πρώτη ε, επίσκεψή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να τον συγχαρώ. Έχει κάνει εξαιρετική εργασία ε, ιδίω ε, έχει γράψει για την Ευρωζώνη και ε, για τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Όσον αφορά τη μελλοντική εργασία και την πορεία της ΕΚΤ ε, είναι υπεύθυνη για την διατήρηση του νομίσματος και την ε, παρουσίαση της πολιτικής και νομίζω ότι η ΕΚΤ θα έπρεπε όντως να, να αυξήσει την ρευστότητα και ιδίω με χρεόγραφα θα μπορέσουν έτσι να ανασάνουν τα κράτη και έτσι θα μπορέσει να εφαρμοστεί μια οικονομική πολιτική η οποία θα υποκινήσει και επενδύσεις. Χρειάζεται βέβαια δημοσιονομική εποπτεία και έλεγχος και πιστεύω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει ε, να παίζει ξιέκτα ένα σημαντικό ρόλο και να συμβάλλει στο να υπάρξει ένα ταμείο το οποίο ε, θα μας ε, ανεξαρτητοποιήσει από τα άλλα ταμεία, δηλαδή να έχουμε ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο. Θα έπρεπε λοιπόν να εξετάσουμε συγχρόνως και τι γενέστε με τα ευρωομόλογα. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος πρέπει να ελεγχθεί και καλό θα είναι όπως είπε ο συνάδελφός μου να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι θα έπρεπε η τράπεζα να δημοσιοποιεί τα έγγραφα τα οποία υποβάλλει στο Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε της Κεντρικής Τραπέζης, σας εύχομαι ε, καλό θάρρος και υπομονή και καλή πορεία. Κυρία Γκάλ Πέλτς, ο κύριος Μπλουμ ε, κινεί μία μπλε κάρτα. Θέλετε να δεχθείτε την ερώτησή του. Έχετε ένα λεπτό κύριε Μπλουμ. Αναφέρατε την αγορά επικινδύνων χρεογράφων. Εγώ είμαι κομμουνιστής και αναρωτιέμαι με ποιου τα χρήματα θα αγοράζετε αυτά τα επικίνδυνα χρεόγραφα. Πού θα βρείτε τα χρήματα από τους συνταξιούχους του Yorkshire, τους δικούς μου ψηφοφόρους, από πού θα χρηματοδοτήσετε αυτό το ίδιο αποτυχημένο πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, ε, δεν συμφωνώ με την ερώτησή σας διότι εσείς ε, ε, κάνετε μία πολύ προκλητική δήλωση για τις περιοχές που πλήττονται από την κρίση. Εάν η ΕΚΤ δεν παίξει το ρόλο που της αρμόζει τότε το ερώτημά σας είναι απλώς διαπίστωση γεγονότων. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ρωτάμε από πού εις βάρος των χρημάτων ποιου θα αγοραστούν αυτά τα επικίνδυνα χρεόγραφα. Θα πρέπει να υπάρξει μια σταθερή οικονομική βάση για να μπορέσει να αντεπεξάλθει η ευρωπαϊκή ζώνη. Ε, αλλά δεν συμμετέχω άρα δεν θέλω να μιλήσω για την καταστροφή του ευρώ. Ευχαριστούμε Ευχαριστώ. κύριε Μπλουμ. επόμενος είναι ο κύριος Χουάνγκοκ Δύο λεπτά παρακαλώ έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η αιτήσια αυτή έκθεση επιτέλους ε, καταρρύπτει κάποια ταμπού. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δηλαδή σκέφτεται ότι μπορεί να πάυσει η αξιολόγηση ή μιλάει για η έκθεση αυτή, για το θετικό Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, να αγοράζει καλυμμένες ομολογίες στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά. Μα έχουμε μία κρίση ρευστότητας μπορεί έτσι να αποφευθεί. Για να πάψει η κρίση του δημόσιου χρέους, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να μπορεί να παρεμβαίνει στις πρωτογενείς αγοράς όταν δεν υπάρχει ρευστότητα. Η ίδια η Γερμανία δυσκολεύεται να βρει χρήματα η έκδοση Ιταλικών ομολόγων γίνεται σε όλο και πιο ψηλά ποσοστά. Δεν υπάρχει παρέμβαση και γι' αυτό το πρόβλημα της Ιταλίας ε, βάζει σε κίνδυνο την υγεία των τραπεζών, οι οποίες δεν δίνουν πιστώσεις και δεν καταφέρνουν να τηρούν τις προδιαγραφές ε, για την ε, ευρωστία τους. Έτσι λοιπόν πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μπορεί όπως και στις Ηνωμένε Πολιτείε να έχει ομόλογα με χαμηλότερα ποσοστά και σε περίπτωση κερδοσκοπίας θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπως γίνεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένε Πολιτείε να εξαγοράζει τα ομόλογα αυτά. Ξέρετε ότι οι χώρε αυτέ χρηματοδοτούνται με πολύ χαμηλά ποσοστά παρά το γεγονό ότι μία από τι δύο χώρε έχει υποβαστεί από τους οίκου αξιολόγηση χρηματοπιστωτική ε, ικανότητας. Θυμόσαστε τη δεκαετία του 20 στη Γερμανία. Η δυνατότητα παραγωγής σήμερα δεν χρησιμοποιείται όπως θα έπρεπε. Δεν υπάρχει ε, πληθωρισμός εξαιτίας της ε, έλψης της ε, ζήτησης. Σήμερα είναι και το κόστος Τη πρώτη ύλη που παίζει ρόλο. Πρέπει επιπλέον, επιπλέον σήμερα να αναγνωρίσουμε ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν αναγνωρίζουν την δημοσιονομική του ορθοδοξία σε περίοδους κρίσης. Ευχαριστώ. Uh, is... Ευχαριστούμε. Η κυρία Στρέτσεκ είναι η επόμενη. 1,5 λεπτό παρακαλώ έχετε στη διάθεσή σας. Ο κύριος Στρέτσεκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Η σημερινή συζήτηση δεν είναι συζήτηση μόνο σημερινή, είναι συζήτηση για το κατά πόσο πρέπει να γίνουν αλλαγέ στη συνθήκη τη Λισαβόνα ή όχι. Είναι συζήτηση για το κατά πόσο χρειαζόμαστε περισσότερη ή λιγότερη ανεξαρτησία τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κατά πόσο χρειαζόμαστε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Πρέπει να απαντηθούν πιο γενικά ερωτήματα δηλαδή σήμερα. Πρόκειται για μια κρίση χρέου ή είναι μια κρίση του ευρώ. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν πρέπει να αναρωτηθούμε το χρέος είναι η αιτία της κρίσης ή το αποτέλεσμα της κρίσης. Ε, το χρέος αυτό που έχει συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια φταίει για την κρίση αυτή ή είναι ε, το χρέος που έχει συσσωρευτεί τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν νομίζω λοιπόν ότι φταίει το ευρώ για την κρίση αυτή. Υπάρχουν διαρθρωτικά ε, προβλήματα εδώ και καιρό στην Ευρωζώνη. Είναι θέμα δημοσιονομικής ευθύνης των κρατών μελών. Όμως, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απαντήσουμε και στο ερώτημα κατά πόσο ο κόσμος είναι διατεθειμένος να αλλάξει τον τρόπο ζωής του, τις προσδοκίες του ή θέλει να συνεχίσει με το κράτος ευημερίας όσο είχε μέχρι τώρα. Υπάρχει μεγάλο βάρος στα δημοσιονομικά μας. Αν δεν απαλλαγούμε από το δημοσιονομικό αυτό βάρος, δεν θα φύγουμε και από την κρίση. Ευχαριστούμε κύριο Μέρφυν. Ο επόμενος, ένα λεπτό παρακαλώ. Έχω εδώ ε, μία, ένα σημείωμα που ε, στάλει στις 5 ε, Αυγούστου ε, το οποίο αναφέρεται σε μέτρα ε, και πλήττουν τους εργαζόμενους και το σημείωμα αυτό υπογράφεται από εσά κύριε Ντράγκη και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αυτό ήταν ε, ένα μέτρο επειδή δεν αγοράζαμε ε, τα Ιταλικά ε, ομόλογα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει συμμετάσχει στην συνωμοσία που έχει πλαϊκή εναντίον της Ελλάδος και της Ιταλίας. Λοιπόν, δεν μπορείτε να μου αποδείξετε ότι είναι ανεξάρτητη η και είναι αντίθετη ή στα συμφέροντα των εργαζομένων υπέρ των, εργαζομένων, υπέρ των συμφερόντων των πλουσίων και διονύζει την κρίση. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Μοργάντη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διακριτικά έπαιξε το ρόλο της αγοράζοντας κρατικά ομόλογα, κρατώντας χαμηλά τον πληθωρισμό, προσπαθώντας να αποτρέψει την οικονομική ύφεση. Δεν σύμφωνο με αυτούς οι οποίοι θέλουν να δώσουν νέε αρμοδιότητες και εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν μπορεί να είναι φέντη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρώπη είναι διαφορετική από τη ΣΥΠΑ. Η Κεντρική Τράπεζα στο μέλλον δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει δημόσια με τις επιστολές της. Θα πρέπει απλά να περιγράφει κάποιους γενικούς στόχους, τους οποίους θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα κράτη-μέλη. Το θέμα του δημοσίου χρέους τέθηκε τους τελευταίους μήνες. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα η οποία έχει πάρα πολλές δυσκολίες λόγω του υψηλού ευρώ να πληρώνει τόσο ακριβά τον δανεισμό της. Θα πρέπει να υπάρξουν λοιπόν ομόλογα ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκά ομόλογα τα οποία να μας βοηθήσουν να αποτρέψουμε την κρίση η οποία έχει αρχίσει. Ο κύριος Παλών έχει δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε Ντράγκη, θα σας καλωσορίσω στην αίθουσα αυτή ως ε, πρόσφατα εκλεγμένου Προέδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής εξ ονόματος της, Ευρωπαϊκής, της Ιταλικής συγγνώμη, αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα σε επίπεδο δημοσιονομικής πειθαρχία. Είναι επίσης σαφές ότι η συζήτηση η οποία γίνεται για τα ευρωομόλογα απαιτούν πάρα πολύ χρόνο και εμείς δεν έχουμε πια χρόνο. Έχουμε άμεσα μέτρα για την ανάπτυξη ενάντια στην ύφεση και στη στασιμότητα. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έπαιξε σημαντικό ρόλο αγοράζοντας ομόλογα κρατών τα οποία είχαν πέσει θύματα κερδοσκοπίας και βοήθησε να μείνει πάρα πολύ χαμηλά ο πληθωρισμός. Έδρασε ταχύτατα και αποτελεσματικά, αλλά η κρίση πλέον έγινε η κρίση του κοινού μας νομίσματος, η κρίση του ευρώ. <clears throat> Αξίζει υποστήριξη όπως και οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. Πρέπει να λειτουργήσει λοιπόν σαν μια πραγματική Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους η Κεντρική Τράπεζα έστω και έμεσα να χρηματοδοτήσει τις χώρες που έχουν ανάγκη έστω και μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έτσι θα πάρει μια θέση πρώτης γραμμής στην αντιμετώπιση της κρίσης του χρέους. Δεν ξέρω βέβαια με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη να περάσουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε μια πραγματικά κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η οποία να είναι οργανισμός εγγυητικός και να έχει τη δυνατότητα να κόβει και χρήμα. Να γίνει ο τελευταίος δανειστής, όπως ακριβώς η Αμερικανική Τράπεζα, να δώσει εγγυήσεις όπως ακριβώς γίνεται με το δολάριο και τη στερλίνα. Αυτό θα βοηθήσει τελικά η Ευρώπη <clears throat> να γίνει μια Ευρώπη αλληλεγγύης και κρατών μελών όπως την ήθελαν ο Αντενάουερ, ο Σπινέλη και ο Ντεγκάσπερη. Uh, Ευχαριστούμε. Ο κύριο Σκυκλούνα τώρα έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Πρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν είναι μόνο κακοτυχία το ότι βρισκόμαστε στην άκρη του γκρεμού. Είναι ένας υπολογισμός που έχει γίνει από όλους τους παράγοντες του ευρώ που μας έφερε στο σημείο αυτό. Είναι μια πρακτική που ακολουθείται για να φτάσει κανείς στο χείλος του γκρεμού, προκειμένου να κερδίσει από τον αντίπαλο. Και αυτό ακριβώς έχουν κάνει ε, οι διάφορες χώρες πιστωτές για να πάρουν από τις πιο δύναμες χώρες όσο μπορούν περισσότερα. Με προγράμματα επίσης λιτότητας, με όρους και προϋποθέσεις και όλα αυτά με τη συνένεση του πληθυσμού με τον ένα τον άλλο τρόπο. Όμως δεν είναι στο συμφέρον της Ευρωζώνης να αφήσει κάποια χώρα να πτωχεύσει. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μάλλον μιλητής, ε, πρέπει να είναι ο δανειστής, ο ίστατος δανειστής, προκειμένου να βρει στο τέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση τις πολιτικές λύσεις που πρέπει. Και όχι να περνάμε ώρες χωρίς λύση. Και με το πακέτο των έξι οδηγιών και με άλλα μέτρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να προχωρήσει σε ευρωμόγολα, να ξεφύγει από τα ταμπού του κουρέματος είναι μια αποστολή σε μια διαδικασία η οποία βέβαια ελοχεύει κινδύνους. Ο κίνδυνος είναι να μείνουμε στην ιστορία σαν μια πολιτική τάξη η οποία με τις στρατηγικές της οδήγησε στην κατάρρευση του ευρώ και την ύφεση. Τεχνικά οι λύσεις είναι γνωστές σε όλους εκείνους που θέλουν να τις ακούσουν. Με όποια μορφή συμπεριλαμβάνουν μέσα τα οποία συνδυάζουν το στοιχείο της αποκοινού ευθύνης όλων των χωρών μελών προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. Οπότε συλλογικά πρέπει να δράσουμε βάσει των αρχών αυτών. Τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες. Πρέπει όμως να δράσουμε και να δράσουμε τώρα πριν να είναι πολύ αργά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τσαρνέκη είναι επόμενος. Δεν είναι όμως εδώ, οπότε έτσι κερδίζουμε χρόνο και δίνω το λόγο στον κύριο Πάσκα. Ένα λεπτό έχετε στη διάθεσή σας, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, διοικητά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 2010, μετά από διαφωνία διαφόρων χωρών, αγόρασε κρατικά ομόλογα στη δευτερογενή αγορά, χωρίς όμως να σταθεροποιηθούν οι αγορές αυτές. Τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι το σύνολο των ομολόγων που αγοράστηκαν είναι τέτοιο που η τράπεζα δεν είναι σε θέση να σταθεροποιήσει το οικονομικό σύστημα. Αν λοιπόν απέτυχε σε αυτό και συνεχίσει να αποτυχαίνει, αυτό σημαίνει ότι διευκολύνεται τελικά η αγορά στην Ευρωζώνη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δηλαδή πρέπει να δείξει μεγαλύτερη ευαισθησία και να στηρίξει το νόμισμά μας περισσότερο και καλύτερα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαγκίνες έχει τώρα το λόγο. Δύο λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την έκθεσή του. Αν και δεν μιλάμε για το 2010 τώρα εδώ, μιλάμε για το μέλλον. Καλωσορίζω τον κύριο Ντράγκη. Το όνομα του προκατόχου σας, του κυρίου Τρασέ, ξέρετε ότι στην Ιρλανδία τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και ελπίζω ότι και το όνομά σας θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο δημοφιλίας. Αν και χθε ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας μου είπε ότι μιλάτε λιγότερο από τον προκάτοχό σας. Ακούσαμε αυτά τα οποία περιμένει κανείς από τη θέση σας. Ήταν ξεκάθαρα αυτά τα οποία είπατε. Και νομίζω ότι τα είπατε με την απαιτούμενη επισημότητα προς όλους μας στην ευκαιρία αυτή. Απαιτείται να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη. Αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο αυτή τη στιγμή σε κλείψη η εμπιστοσύνη. Βλέπω εδώ τον κύριο Μπλουμ, ο οποίος έθεσε αρκετές ερωτήσεις και πάντα θέτει ερωτήσεις όπως πρέπει στη δημοκρατία και θα ήθελα να του πω να προσέχει το τι εύχεται. Αυτό το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα της Ένωσης, δεν είναι πρόβλημα της Ευρωζώνης. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι σφαιρικό πρόβλημα, είναι συνολικό πρόβλημα. Και αν πράγματι αποτύχει το ευρώ, διαλυθεί το ευρώ και αν καταργηθεί το κοινοβούλιο, τότε κύριε Μπλουμ και η δική σας χώρα θα αντιμετωπίσει απίστευτα προβλήματα. Θα ήθελα λοιπόν στις συζητήσεις που γίνονται εν θερμό να αναγνωρίσουμε τη σημασία αυτών που λέμε και το βάρος των λέξεών μας στην προσπάθεια αποκατάστασης εμπιστοσύνης. Μιλάμε για ανθρώπους τους οποίους αντιπροσωπεύουμε και οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτοί που είναι οι αντιπρόσωποι τους και που είναι στην εξουσία ε, θα πρέπει να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει. Φυσικά και θα δεχθώ ερωτήσεις, περιμένετε όμως πρώτα να τελειώσω, λέει η κυρία Μαγκίνες. Το θέμα δεν είναι να βλέπουμε τι έγινε στο παρελθόν. Το πρόβλημα σήμερα είναι παγκόσμιο, είναι μεγάλο για όλους. Απαιτείται να πετύχει η κυρία το ευρώ και απαιτείται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να είναι ένα σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας αποκατάστασης της εμπιστοσύνης και των νέων μέτρων τα οποία θα απαιτηθούν στο μέλλον. Συγγνώμη γιατί ε, μίλησα περισσότερο. Νομίζω ότι είχατε κάποια αιτιολογία. Ο κύριος Μπλουμ έχει μία μπλε κάρτα, το έχετε δεκτεί και ο κύριος Μίτσελ έχει μία μπλε κάρτα. Δέχεστε και αυτήν. Είναι άλλο ένα λεπτό. Λοιπόν κύριε Μπλουμ μισό λεπτό. Ε, δεν είπα ότι θέλω να αποτύχει, αλλά υπάρχει το συνέστημα στο Ευρωκοινοβούλιο ότι μας έχει πλήξει ένα τσουνάμι ή ένας αστεροειδής, ότι είναι κάτι για το οποίο δεν φταίμε εμείς. Ε, Υπάρχει όμως μία κατάσταση την οποία εμείς δημιουργήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι θεομηνία, είναι κάτι το οποίο εμείς προκαλέσαμε. Δεν νομίζω ότι αυτό ήταν ερώτηση, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Μαγκίνες. Ε, εγώ είμαι ήρεμη. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά αυτό απαιτεί εφόσον δημιουργήσαμε το πρόβλημα συλλογικά να το λύσουμε, διότι φωνάζοντας ε, και εξαπτώμενοι δεν θα το λύσουμε και δεν θα μας ακούει και κανείς. Ε, ευχαριστώ για τη σύντομη απάντηση. Κύριε Μίτσελ, έχετε το λόγο. Δεν ξέρω αν η κυρία Μαγκίνε συμφωνεί μαζί μου δεδομένη στις εμπειρίες που είχαμε στην Ιρλανδία με τους οικονομικούς σχολιαστές ε, όταν ήταν στην εχμή το πρόβλημα ε, ε, ότι η συμπεριφορά ήταν απαράδεκτη. Κυρία Μαγκίνες για μισό λεπτό πρέπει κάτι να πω ότι είμαι οικονομολόγος ε, στα θέματα γεωργίας πρέπει να πω και είμαι, αντιμετωπίζω πολύ σοβαρά το ερώτημα του κυρίου Μίτσελ και πιστεύω ότι όποιος εμπλέκεται σε αυτή τη συζήτηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις των σχολείων του διότι μπορεί η, η, ε, κυβέρνηση ε, να ε, ε, μπορεί άλλοι να μπορούν να αποχωρήσουν αλλά εμείς πρέπει να χρησιμοποιούμε όρους οι οποίοι έχουν νόημα και να ακολουθούμε με πράξη τα λόγια μας. Ε, ευχαριστώ. Είσαστε τόσο προκλητικοί ώστε ο κύριο Ρούμπικ επισύει την μπλε κάρτα. Δέχεστε την μπλε κάρτα του κυρίου Ρούμπικ γιατί νομίζω ότι θα είναι η τελευταία. Κύριε Ρούμπικ μισό λεπτό. Θέλω να ευχαριστήσω γιατί για ορισμένους καλύτερα θα ήταν προσωπικά να έχουν ένα δικό τους νόμισμα και να ξοδεύουν τα δικά τους ε, χρήματα. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν και άρα θα πρέπει στις χρηματαγορές τώρα να φροντίσουμε να συνεχιστεί να υπάρξει ρευστότητα και θέλω να ρωτήσω την κυρία Μαγκίνες αυτό που έγινε εχθές όταν ε, κεντρικές τράπεζες ε, έριξαν χρήματα στις αγορές μαζικά θα βοηθήσει ή θα υπάρξει ένα double dip. Ήδη έχει γίνει αυτό, ανάλογα με το μήνυμα το οποίο θέλουμε να στείλουμε για να υπερασπιστούμε το σύστημα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να θεωρηθούμε σαν έθνος αν θέλετε συνολικά. Και όπως είπε και ο κύριο Βαν Ρομπόι, μια οικονομική αλλαγή γίνεται με ένα κλικ στο ποντίκι στον υπολογιστή, ενώ μια πολιτική αλλαγή απαιτεί προετοιμασία, απαιτεί χρόνο. Θα το πετύχουμε όμως, χρειάζεται όμως να είμαστε συντονισμένοι και αποφασιστικοί. Σας ευχαριστώ κυρία Μαγκίνες. Ε, απλά σα απειλούσα, δεν σα πέταγα το σφυρί, λέει ο Πρόεδρο. Η κυρία Ποδηματά, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με την ε, έκθεση του κυρίου Τρεμόζα η Μπαλσέη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει πληρω κύριε Πρόεδρε, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει παίξει ενεργό και αποφασιστικό ρόλο σε όλη τη διάρκεια της κρίσης, αφότου ξεκίνησαν οι αναταραχές στις χρηματοπιστωτικές αγορές το 2007, το 2008 μέχρι βεβαίω τι παρεμβάσει στι δευτερογενεί αγορέ των τίτλων δημοσίου χρέου τη ευρωζώνη. παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε και γνωρίζετε ότι η κρίση εξελίχθηκε δεν περιορίστηκε και έχει πάρει πλέον συστημικό χαρακτήρα και βεβαίω είναι προφανέ ότι αυτό δεν αποτελεί ευθύνη τη ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα όπω συστηματικά και κατ' επανάληψη έχει επισημάνει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο η διεύρυνση και η διάχυση της κρίσης είναι αποτέλεσμα της διστακτικότητας της αναποφασιστικότητας και των καθυστερήσεων στη λήψη και στην εφαρμογή των κατάλληλων αποφάσεων πρωτίστως σε πολιτικό επίπεδο από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. κύριε πρόεδρε η χθεσινή απόφαση της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας στην οποία αναφερθήκατε να συντονίσει τις κινήσεις της με τις πέντε μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο για να αυξήσουν τη ρευστότητα στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει αναμφισβήτητα μια θετική διάσταση ε, είναι μια απόφαση που θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα προσωρινά. γνωρίζουμε όλοι ότι χρειάζεται άμεσα μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική απάντηση στην κρίση που θα πηγαίνει πιο πέρα και θα συνδυάζεται με τους κανόνες της αυστηρότερης δημοσιονομικής πειθαρχίας στους οποίους αναφερθήκατε με το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο όπως το χαρακτηρίσατε. κύριε πρόεδρε το είπαν και άλλοι συνάδελφοι σεβόμαστε απολύτως την ανεξαρτησία της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας η οποία ωστόσο πέρα από τη σταθερότητα των τιμών είναι ο θεματοφύλακας του ευρώ του κοινού νομίσματος και πρωτίστως αυτό το ρόλο καλείται σήμερα εκτάκτως να παίξει. γνωρίζετε και γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει τρόπος να βγούμε από την κρίση Χωρί ενισχυμένο ρόλο της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας. επαφίεται βεβαίω σε εσά και στο εκτελεστικό συμβούλιο της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας να εξετάσετε όλες τις προτάσεις και να αποφασίσετε το πώς. ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Uh, ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, να πω ότι θα δώσω σε τρία μέλη το λόγο στα πλαίσια του ΚΑΤΣΤΙΑΙ, Μάλλο, Φερέρα και Ντερόσα. Ενημερωτικά σας το είπα αυτό. Ο κύριος Λούντβικσον έχει λοιπόν το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχει μεγάλη σημασία να παρατηρήσει κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη διάρκεια της ευρωκρίσης εισαγωγικά έχει κάνει μια καλή δουλειά, μια καλή προσπάθεια. Και στον τομέα των επιτοκίων έχουμε φτάσει σε ένα αρκετά χαμηλό, ανεκτά χαμηλό επίπεδο. Η υποστήριξη ε, των ομολόγων ε, φυσικά των ασθενών χωρών είναι κάτι το οποίο χρήζει περισσότερη ισορρόπησης. Το θέμα είναι να έχουμε στη διάθεσή μας ένα πραγματικό μέσο, ένα σύνολο μέσων, ένα toolbox το οποίο να μας βοηθήσει να δούμε ποια είναι η κρίση. Δεν έχει τελειώσει η κρίση σε καμία περίπτωση. Και γι' αυτό έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σήμερα που αμφισβητείται το σύνολο των μορφών συνεργασίας μας. Ένα μη αναμενόμενο σοκ μπορεί λοιπόν να δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα και στις κυρίαρχες χώρες. Ένα Lehman Brothers 2 είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί ξανά και ξανά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει σαν πολιτικοί να προσπαθήσουμε να το αποτρέψουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι καμία από τις, ή κάποιες από τις λύσεις θα πρέπει να εμπλέκουν και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί έτσι Θα πρέπει οι τράπεζες να μπορέσουν σαν γι' αυτοί, να μπορέσουν να λειτουργήσουν σαν δανειστής τελευταίας ευκαιρίας αν θέλετε. Αυτό είναι απαραίτητο μέσο πρόθεσμα και μάκρο πρόθεσμα μια πιο ε, προληπτική πολιτική θα αποτρέψει βέβαια τους κινδύνους σε επίπεδο προϋπολογισμών κρατών μελών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να επιδιώξουμε. Θα πρέπει όμως να το επιδιώξουμε ισορροπώντας το και με άλλους κινδύνους οι οποίοι απειλούν τις διάφορες χώρες. Πρέπει λοιπόν να ξανασκεφτούμε τον τρόπο λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να μπορέσει η τράπεζα να κάνει περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία επιτελεί σήμερα. Μόνο τότε θα ξεφύγουμε από τις αναταράξεις και τα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν τώρα. Δεν έχει νόημα να περιμένουμε ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ όλους. Thank you. Ε, Ευχαριστούμε. Catch the eye. Ο κύριος Μάουρο είναι ο πρώτος. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως καταλάβατε από τις παρεμβάσεις των περισσότερων συναδέλφων, παραδόξως σήμερα κανένας δεν ζητά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ξεφύγει από τις αρμοδιότητές της. Όλοι εκφράζουμε ευχές σε επίπεδο οράματος. Μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα πάντα βέβαια με τα ίδια αυτής χαρακτηριστικά και με την ίδια της τη φύση αλλά είναι σαφές ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε, γιατί είναι επίσης προφανές ότι τη στιγμή κατά την οποία ε, θεωρήσετε ότι η πρόταση του κυρίου Τρεμόσα είναι επαρκής, είναι ενδιαφέρουσα και θα λειτουργήσει θετικά, τότε θα δώσουμε τη δυνατότητα στους πολιτικούς να μας οδηγήσουν εκτός προβλήματος. Λοιπόν, εδώ η αναποφασιστικότητα είναι μοιραία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε την σύγκρουση η οποία σοβεί στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία μας απαγορεύει να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Είμαστε πολλοί που θέλουμε να υπάρξουν συγκροτημένες αλλαγές για να βοηθηθεί η Ευρώπη να συνεχίσει και να πετύχει. Ευχαριστώ. Η κυρία Φερέιρα, ένα λεπτό. Καλώς ήρθατε στο κοινοβούλιο μας κύριε Ντράγκη. Βιώνουμε δραματικές στιγμές, βιώνουμε δύσκολες στιγμές. Απαιτείται να υπάρξει μια επίγουσα και δραματική θα έλεγα αντίδραση, μια αντίδραση δραματική η οποία να σπάσει αυτό το φαύλο κύκλο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και οι χώρες. Θα πρέπει να μην καταστραφεί από τις υπηρεσίες αξιολόγησης και από τους κερδοσκόπους το νόμισμά μας στην έκθεση σε Αυτό το οποίο γίνεται είναι να προτείνονται μέτρα έτσι ώστε να δημιουργηθεί ουσιαστικά ένα Ευρωπαϊκό Οικονομικό Υπουργείο. Όλα αυτά είναι καλά θεωρητικά. Τώρα βιαζόμαστε, σήμερα βιαζόμαστε. Τι έχουμε στα χέρια μας, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τεχνικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γνωρίζει το τι είναι απαραίτητο να συμβεί. Δεν πρέπει να φοβάστε να πάρετε μέτρα κύριε Ντράγκη. Δεν πρέπει να φοβάστε να δράσετε λόγω κάποιων πάρα πολύ περιοριστικών ερμηνεών της εντολής την οποία έχετε σαν τράπεζα. Πρέπει να κάνετε ό,τι μπορείτε για να σώσετε το ευρώ. Αυτό περιμένουν οι πολίτες από σας κύριε Ντράγκη. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο στα πλαίσια του ΚΑΤΣΔΙ ε, είναι ο κύριος Ντερόσα για ένα λεπτό. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Ντράγκη. Πράγματι χρειάζεται μεγαλύτερη παρέμβαση της ΕΚΤ. Αλλά οι πολίτες δεν θα δεχθούν αυτή την παρέμβαση αν δεν υπάρξει μεγαλύτερος δημοκρατικός έλεγχος και κοινωνική δικαιοσύνη. Τότε μόνο θα δεχθούν τις παρεμβάσεις μας. Για να αποφύγουμε την πτώση ε, στη δεκαετία του 30 θα πρέπει να σώσουμε το ευρώ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να γίνει ο δανειστής της τελευταίας ευκαιρίας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος για να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτά τα οποία προτείνονται για σχέση ΑΕΠ και χρέους 25% πολύ πιο χαμηλά από το 60% είναι σίγουρα δύσκολα να γίνεται. Στην ουσία εμείς έχουμε εθνικοποιήσει το ιδιωτικό χρέος των τραπεζών. Στις, ε, τα χρέη των γερμανικών, των γαλλικών τραπεζών τα έχουμε αναλάβει εμείς σαν κράτη. Δεν μπορούμε όμως να τα καταφέρουμε, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε το χρέος αυτό εφόσον μένουμε πάντα στην, στενά, στην στενή εντολή της δημοσιονομικής πειθαρχίας και συστολής. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Απαιτείται ανάπτυξη στην Ευρώπη, απαιτούνται ευρωομόλογα και κυρίως απαιτείται αλληλεγγύη. Uh, Ευχαριστούμε. Έτσι ολοκληρώνεται η παρουσία των ομιλιών. Ο κύριος Δράκη θα έχει το λόγο τώρα και σας εύχομαι και εγώ κάθε επιτυχία στο τόσο δύσκολο έργο που έχετε μπροστά σας. Παρακαλώ. President. Thanks. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις δηλώσεις τους, τις ε, συμβολές τους και θα ήθελα να πω από την αρχή ότι προσβλέπω εις ε, την ανταλλαγή απόψεων και στις ευκαιρίες που θα έχουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις, να σκεφτούμε από κοινού ε, και να αντιμετωπίσουμε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία νομίζω ότι πολλές από τις δηλώσεις του σου περιλαμβάνονται σε ένα κεφάλαιο. Πώς θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την ε, εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη. Και αυτή η διαδικασία θα χρειαστεί να βασιστεί σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι αυτό το οποίο ε, θεωρώ σαν ένα γυροβόλιο μακροπρόθεσμα, δηλαδή ε, μία αναμόρφωση των φορολογικών κανόνων βάσει μια συμφωνίας επί νέων φορολογικών προτύπων ε, ε, κανόνων για να μπορέσει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ή στην Ευρωζώνη. Αυτός ε, ο σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα μας πούν εάν ε, έχουμε προχωρήσει ή όχι αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι αποκαθιστά την εμπιστοσύνη μακροπρόθεσμα και αυτό είναι αναγκαίο για να λειτουργήσουν οι δύο άλλοι πυλώνες δηλαδή για να μπορέσουν ε, να ε, ε, προχωρήσουν ο μηχανισμός σταθερότητος στην Ευρωζώνη το EFSF το οποίο χρειάζεται ακόμη ορισμένες τελειοποιήσεις και τέλος η αντίδραση στην οικονομική πολιτική και στον τομέα αυτό έχουμε προχωρήσει πολύ διότι όπως σας είπα πιστεύω ότι τα κράτη τώρα έχουν εφικραμιστεί παρόλο που βλέπουμε ε, με ένα βίωνο μέλλον αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ε, πόσο θα εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες προτείνονται και δεν πρέπει να εστιαστούν μόνο σε δημοσιονομικά θέματα αλλά θα χρειαστούν και διαρθρωτικές αλλαγές που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες επί των οποίων μπορούμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη. Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΚΤ σε ο σύνολο αυτό. Ορισμένοι έθεσαν το ερώτημα. Άλλοι είπαν πρέπει να κάνει περισσότερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλοι είπαν πρέπει να κάνει λιγότερα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όμως μπορεί να λειτουργήσει στα πλαίσια της συνθήκης. Δεν μπορεί λοιπόν να τη ζητηθεί να κάνει πράγματα τα οποία υπερβαίνουν την ε, ε, συνθήκη. Είναι ο δανειοδότης τελευταίας διαφυγής ε, για ε, τις χρεγωμένες ε, χώρες και βλέπουμε τώρα ότι το θέμα δεν είναι το ποσό της ρευστότητος αλλά το να κυκλοφορεί αυτή η ρευστότητα μέσω του τραπεζικού συστήματος, μέσω των οικονομικών και πιστοληπτικών συστημάτων και ε, πρέπει ε, να αποκαταστήσουμε ε, τις πιστοτικές διόδους κατά τρόπον ώστε να ενδυναμώσουμε την οικονομία και τα ευρωπαϊκά χρηματοοικονομικά Ινστιτούτα που χρειάζονται βοήθεια. Γενικώ θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα πρόσβαση ε, των ε, ε, κρατών στις αγορές και δεν χρειάζονται τις τράπεζες αλλά το σύστημα αρχίζει να βελτιώνεται παρόλο που βλέπουμε μεγάλη στην ενότητα πιστοτική τελευταίως και αυτό βεβαίως επηρεάζει δυσμενώς τις επιχειρήσεις για τους επόμενους μήνες. Ορισμένοι αναφέρθηκα στο SMP, ε, το πρόγραμμα για την αγορά χρεογράφων. Πρέπει να σας πω όπως έχω ήδη πει στο παρελθόν για να λειτουργήσει το πρόγραμμα αυτό πρέπει να έχετε εξασφαλίσει ότι μπορεί να έχουν αποκατασταθεί ε, τα ε, κανάλια μεταδόσεως χρηματοοικονομικής πολιτικής. Πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η μεταφορά των ε, χρηματικών πόρων και αυτό έχουμε προσπαθήσει. Είναι ένα άτυπο μέτρο και ως εκ τούτου θα είναι ένα προσωρινό περιορισμένο μέτρο και θα σας πω τι εννοώ για περιορισμένο δεν είναι ούτε ατέρμον ούτε αιώνιο και η ΕΚΤ μπορεί να λειτουργήσει μόνο στα πλαίσια της συνθήκης. Θα ήταν λάθος να κινηθεί η ΕΚΤ εκτός της συνθήκης και θα ήταν επίσης λανθασμένο να το απαιτήσουμε διότι έτσι θα υποθάλπαμε την αξιοπιστία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία αυτή τη στιγμή είναι η πιο ισχυρή υπογραφή στην Ευρωζώνη, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη. Θέλω λοιπόν ε, να επαναλάβω αυτά που ελέγχθησαν σχετικά με την επικοινωνία ε, διότι ιδίω σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση ακραίων δυσχεριών δεν έχει νόημα να υπάρχει μια κακοφωνία και διάφοροι να προκαταλαμβάνουν το τι πρόκειται να συμβεί σύμφωνα με το δικό του σκεπτικό και να παρουσιάζουν τις δικές τους απόψεις αντί για την συλλογική παρουσίαση. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να μεταφέρω και στα υπόλοιπα μέτρα του Συμβουλίου Διακυβέρνησης. Θα προσπαθήσω λοιπόν να συνεχίσω τις προσπάθειές μου. Προσβλέπω στην επόμενη συνάντησή μας σε λίγες μέρες στην Επιτροπή Οικονομικών και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ. Πρόεδρε. Πρόεδρε. Για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, στρέφομαι στον εισηγητή, τον κύριο Τρεμόσα. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για όσα είπατε στη συζήτηση αυτή. Κύριε Ντράγκη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δραστικά παρέμβει και έχει αποφύγει μεγαλύτερη καταστροφή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έσωσε πολλούς Ευρωπαίους από το να ζήσουν ε, ε, μαζική τραπεζική καταστροφή. Οι οικονομικές αγορές δεν δείχνουν εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη ως μια Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Όμως η πίεση των αγορών μπορεί και να βοηθήσει να υποχρέωσουμε τις πιο δύναμες χώρε να περιορίσουν τον προπολογισμό τους και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά του. Η κρίση αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για περισσότερη δημοσιονομική ένωση μέσα στην ε, Ευρωπαϊκή, μέσα στην Ευρωζώνη και μπορούν έτσι να χάσουν ένα μέρος της κυριαρχίας τους στα κράτη-μέλη. Η ευρωπαϊκή κρίση είναι όμως και μια πολιτική κρίση. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ανακάλυψαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τα δικά της μέσα για να δράσει σε περίπτωση τέτοιας μεγάλης κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τους δικούς της πόρους για να αναπτύξει τη δικιά της πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδείχθηκε αδύναμη, ε, χωρίς ε, δημοκρατική νομιμότητα, όπως είπε κάποιος εδώ. Κύριε Ντράκη, καλή επιτυχία στο έργο σας περισσότερο από ποτέ λέμε έχουμε εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ πολύ. Thank uh, Καλώς, έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση για το θέμα αυτό που ήταν η ετήσια έκθεση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα ψηφίσουμε την έκθεση